Συνάδελφοι, ε, ξεκινάμε. Είχαμε τη συνεδρία των συντονιστών. Και τώρα θα προχωρήσουμε, θα συνεδριάσουμε εκ νέου μέχρι τις 5.30. Στις 5.30 θα έχουμε την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν έχουμε και, τις, και τη γεωργίες. Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο, οπότε πάμε στο 12 κατευθείαν για τα ενετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο του 2014. Εμείς έχουμε να συντάξουμε γνωμοδότηση ο δικός μας εισηγητής ε, είναι ο κύριος Φρουντσούλικα και έχετε το λόγο παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προσπάθησα να καλύψω στο δυνατόν περισσότερα θέματα κατά τη σύνταξη της ονομοδότησης για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε στεναρά τη θέση μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πιστεύω ότι πρέπει να αναδείξουμε τη σύνδεση που έχει η σχεδιασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταπολέμηση της φτώχειας, η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, η καλή διακυβέρνηση και η ασφάλεια και ελευθερία. Κύριε. Ο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης και με αυτόν στο λόγο θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων στις διάφορες χώρες του κόσμου. Γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί προς, τη, προς αυτόν τον σκοπό είναι τα κατάλληλα, διευκολύνουν και το έργο της και το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Πρέπει να ενισχύσουμε την ιδέα της λογοδοσίας και επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι αν σωστά εφαρμοστεί αυτή η λογοδοσία δεν ε, δημιουργεί προβλήματα στην ευρωπαϊκή οικονομία, κάθε άλλο μας βοηθάει να επιτύχουμε και τους κοινωνικούς και τους οικονομικούς και τους περιβαλλοντικούς μας στόχους και εντός των σύνορων της Ευρώπης και εκτός. Ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Ένας λόγος παραπάνω να εστιάσουμε στα γεννησιουργά αίτια αυτών των ροών, των μεταναστευτικών ροών, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προβλήματα ασφαλείας, είναι προβλήματα στο περιβάλλον, είναι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατάρρευση του κράτους δικαίου δεν είναι διαπραγματεύσιμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδες ελευθερίες στο πλαίσιο του πολιτικού δηλαδή λόγω με τρίτες χώρες. Στο κείμενό μου αναφέρομαι επίσης στην σημασία που έχει η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια αναπτυξιακής συνεργασίας να περνάει μέσα από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ε, τοπικές έτσι ώστε να πιάνουν ε, τόπο τα χρήματα της Ένωσης. Σήμερα το πρωί είχαμε συνάντηση της ομάδας εργασίας Α και συζητούσαμε για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο έχει υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση διάφορες χώρες. Σήμερα συζητήσαμε τη Μαγαδασκάρη. Πρέπει να ξεκαθαρίζουμε προς όλες εκείνες τις κυβερνήσεις τις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ο σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων, των συγκαλιστικών δικαιωμάτων ε, και η καταπολέμηση της διαφθοράς, όλα αυτά είναι διαπραγματεύτα. Στις συμφωνίες με χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο, τις οποίες συνάπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ε, σαφείς ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στις εμπορικές συμφωνίες, συμφωνίες, συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας. Πρέπει επίσης να τονίσουμε το ρόλο που έχει η χρήση της, της βοήθειας αναπτυξιακής συνεργασίας για την πρόθεση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αυτά κυρία σημεία που ήθελα, στα οποία εγώ θέλω να σταθώ. Ευχαριστώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας και να απαντήσω σε τυχόν απορίες ή άλλα σχόλια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πρέντα, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Φρουντζουλίκα για τη γνωμοδότησή του. Ως εισηγητής για αυτό το θέμα στην Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι και συνέταξα τη δική μου έκθεση, ε, όπου τονίζω τη σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη, εφόσον βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Το κείμενό μου είναι σύντομο, δεν είναι κατάλογος όλων των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε επέλεξα ένα σύντομο κείμενο που προσπαθώ να εστιάσω την προσοχή στα πιο σημαντικά θέματα. Τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ώστε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις σχέσεις μας με τις ε, τρίτες χώρες. Δεν ήθελα λοιπόν να κάνω έναν ολόκληρο κατάλογο όλων των παραβιάσεων, όπως έλεγα. Συνέταξα την έκθεσή μου εξετάζοντα τα μέσα της Ευρωπαϊκή Ένωσης στις σχέσεις της με τι τρίτε χώρε, του διαλόγου, για παράδειγμα, που έχουμε με τρίτε χώρε για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι κατευθυντήριες γραμμέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το πρόγραμμα Δράση της Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Οπότε ανέλησα όλα αυτά τα μέσα, ό, όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και εστίασα σε αυτούς τους βασικούς άξονες, δηλαδή δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Επέμεινα για ε, θέματα δημοκρατίας, διότι τελευταία έχουμε αφιερώσει λιγότερη προσοχή <clears throat> στο θέμα της εδραίωσης της δημοκρατίας και ε, την σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία δεν μπορούμε να στηρίξουμε και να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς δημοκρατία. Γι' αυτό και επέμεινα σε αυτό το συσχετισμό. Ένα από τα κύρια θέματα, μάλλον μηνύματα της εκθεσής μου, που είναι επίσης ε, ε, επίκαιρο για την σημερινή συζήτηση εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης, είναι ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τις πολιτικές μας με τρόπο ώστε να εδρεωθεί, να παγιωθεί η δημοκρατία και να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλώ δηλαδή για την εμπορική πολιτική, για την αναπτυξιακή πολιτική, αλλά και για την πολιτική γυτνίασης και διεύρυνσης. Όλες αυτές οι πολιτικές μπορούν να συμβάλλουν, δύνανται να συμβάλλουν μάλλον, σε στην πρόθεση της δημοκρατίας και στην, ε, ε, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που με την ανάπτυξη, της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ανέφερα την ε, ατζέντα του 2030 ούτε τους νέους στόχους γιατί τότε δεν είχαμε καταλήξει ακόμα σε αυτούς. Επίσης υπευλήθησαν τροπολογίες στη συνέχεια ώστε να ληφθεί υπόψη η καινούρια ατζέντα, η πρόσφατη, καθώς και οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης επέμεινα για τη σχέση ανάμεσα στην συνοχή μάλλον ε, στη συνοχή για τέτοια θέματα, ε, καθώς ε, την χάνω να είμαι εισηγητής για αυτό το θέμα εδώ στην ΔΕΒΕ, και μια άλλη προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ η σχέση αυτή θα πρέπει να συγκεντρώνει την προσοχή μας. Προσβλέπω λοιπόν στη συμβολή της Επιτροπής ΔΕΒΕ μέσω της ε, γνωμοδότησης του κυρίου Φρουντζουλίκα έτσι θα μπορέσουμε να συνομιλούμε και στην ε, μητρική μας γλώσσα, πράγμα που δεν μας συμβαίνει πολύ συχνά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν ήμασταν ε, στη Νέα Υόρκη για τα SDG, τους στόχους, είχαμε μια σημαντική ενδιαφέρουσα συνεδρίαση με ταξί στατιστικολόγων. Ξέρετε πως έχουν 19 στόχους και μετά 169 υποστόχους. Θα αναπτυχθούν και στόχοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση. Θα ήταν ίσως λοιπόν ενδιαφέρον να συμπληρωθεί. Αυτή, αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Τώρα να δούμε αν αυτό θα χρησιμεύσει και ως εργαλείο για την Ένωση για να εξετάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν και νομίζω πως ε, έχετε δίκιο που λέτε ότι δεν πρέπει να κάνουμε καταλόγους με όλα, γιατί ο κίνδυνος είναι να μην κάνουμε τίποτα τελικά, να αλλάζουμε ε, τα πράγματα. Ο στόχος είναι να αλλάξουν τα πράγματα και όχι να κάνουμε, να κάνουμε καταλόγους. Η Μπέτρις έχει ζητήσει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να, σας να ευχαριστήσω τον κύριο Φρουντσουλίκα για την έκθεσή του και για το κείμενο αυτό. Πιστεύω ότι είναι αρκετά συμπυκνωμένο αλλά ταυτόχρονα ε, επεξηγηματικό για το τι μπορεί να είναι μια γνωμοδότηση της ΔΕΒΕ για αυτή την έκθεση του κυρίου Πρέντα. Μου άρεσε πολύ που δεν ά. Ε, που, που τονίζει τη δημοκρατία ως βάση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο κύριος Πρέντα στην έκθεσή του και πιστεύω πως μέσω αυτής εδώ της νομοδότησης μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο αυτή την ιδέα ότι δηλαδή η εδραίωση, η παγίωση της δημοκρατίας που αποτελεί το θεμέλιο της ειρήνης και της δικαιοσύνης μέσω ισχυρών θεσμών είναι αλήθεια και έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα γιατί τώρα ένας από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης το αναφέρει ρητά αυτό. Είναι μια από τις μεγάλες προόδους ε, της ατζέντα για την βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030 και μέσα στα σχόλια και τη μικρή συμβολή που θέλω εγώ να προσφέρω στον κύριο Φουντζουλίτσα ε, είναι ακριβώς αυτό το να τονίσουμε ότι υπάρχει αυτός ο στόχος για την ε, ρητή βιώσιμη ανάπτυξη, για το στόχο 16 μέσα στο πλαίσιο της ατζέντα των στόχων για το 2032 και όπως έλεγε και η Λίντα τώρα, οι δείκτες οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν και μια μέτρηση της υλοποίησης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των σχετικών προδιαγραφών. Ταυτόχρονα θα ήθελα να τονίσω ότι ενώ εξακολουθούμε να είμαστε η αναφορά για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είμαστε τόσο εντάξει όταν εμείς πρέπει να τηρήσουμε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο αυστηροί είμαστε με τις άλλες χώρες. Ε, δηλαδή θα πρέπει και αυτό να το αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται δηλαδή πιο αποτελεσματική χρήση ε, και πιο αποφασιστική χρήση των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο 4 συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη γνωμοδότηση που, κάνουμε, δηλαδή να, να κάνουμε, να φτιάξουμε μάλλον το αίτημα που κάνουμε προς την Κομισιόν για να φτιάξουμε ένα διεθνές μέσο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αυτήν εδώ την έκθεση θα έπρεπε ίσως να το αναφέρουμε. Έχω να κάνω μια πρόταση ότι δηλαδή θα είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε αυτή την πτυχή της δέσμευσης του υποχρεωτικού χαρακτήρα των ε, επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι κάτι που ήδη οι επιχειρήσει μα θέλουν να κάνουν. Δηλαδή πολλέ φορέ μιλάμε για δεσμευτικέ υποχρεώσει, λε και ήταν κάτι που εμεί επιβάλλουμε ω τιμωρία κατά κάποιο τρόπο. Ενώ τελικά οι ίδιε οι επιχειρήσει θέλουν να συμπεριφερθούν σωστά και να αποτελούν το παράδειγμα για το πώ κανεί πρέπει να συμπεριφερθεί ώστε να είναι στο επίπεδο που πρέπει για να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του. Γι' Και αυτό είναι ένα σπουδαίο μέτρο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σωστό ε, δρόμο. Επιπλέον έχω κάποια σχόλια όσον αφορά τις πτυχές αύξησης της διαφάνειας ε, στα αναπτυξιακά θέματα. Τα προγράμματα δηλαδή ε, τα αναπτυξιακά να, έχουν, να περιλαμβάνουν μια ρήτρα που να αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε τόσο σύντομη βέβαια γνωμοδότηση και τόσο συνοπτική, θα μπορούσαμε ίσως εδώ να τονίσουμε περισσότερο στο τελευταίο σημείο τα θέματα της βίας κατά των γυναικών και ίσως να μιλήσουμε και για την ε, διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης που είναι δεσμευτική και που η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υπογράψει και κυρώσει. Ευχαριστώ. Μαρία Χόιμπρουκ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντάκτη της γνωμοδότησης. Θα ήθελα όμως να προτείνω και κάποιες προσθήκες και κάποιες τροποποίησεις δίνεται έμφαση ε, ανάμεσα στα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για τον προβεώθηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων αναφέρεστε στην πολιτική για την ανάπτυξη της Ένωσης και τις ρήτες τρεις ανθρωπινών δικαιωμάτων που μπορούν να ε, αναφερθούν. Ή επίσης λέτε ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα για το κοινωνικά δικαιώματα και το εργατικό δίκαιο στις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Αυτά είναι πιστεύω κατά την άποψή μου στοιχεία που πρέπει να τονιστούν στην έκθεση. Επίσης να τονίσουμε το ζήτημα του δικαιώματος στην υγεία και επίσης το δικαιώματος στα αναπαραγωγικά δικαιώματα. είναι ένας τομέας στον οποίο ε, δεν έχουμε πάει όσο μακριά θα έπρεπε να έχουμε ε, υιοθετήσει μια συνεκτική πολιτική σε αυτόν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, γνωμοδότηση αυτή. <clears throat> Θεωρούμε ότι αποτελεί μια πολύ καλή βάση θα θέλαμε όμως να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις που πιστεύουμε ότι θα εμπλούτιζαν αυτή τη γνωμοδότηση. Μία είναι ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι το μοναδικό μέσο απέναντι σε κατάσταση φτώχειας ή κατά ε, πάτησης δικαιωμάτων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι αναπτυξιακές πολιτικές, αλλά υπάρχει και ανάγκη να κινηθούμε από μια βοήθεια αναπτυξιακή σε μια πολιτική δίκαιη, γενική, σφαιρική, που θα έχει τη δυνατότητα να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις στην καθημερινή ζωή του κόσμου. Γιατί η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι ατμοσφαιρικό, περιβαλλοντικό ή μετεωρολογικό φαινόμενο από το οποίο είναι αναποφευκτό. Έχει ωστόσο πολύ σημαντικέ πολιτικέ συνέπειε αλλά και οικονομικέ συνέπειε. Και για να μπορέσουμε να, ε, να χτυπήσουμε στη ρίζα το, το κακό για τι στόχε, Ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε ποιες είναι οι στρεβλές επιπτώσεις ας πούμε της εμπορικής πολιτικής. Ε, οι επιχειρήσεις μας δεν θα πρέπει να πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες όπως βλέπουμε να γίνεται καθημερινά πολλές φορές. Επίσης ε, υποστηρίζουμε την δέσμευση όσον αφορά την εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί μιλάμε για ρυθμίσεις όπως ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τους στόχους της, ανα... της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε... Θα πρέπει να έχουμε πλαίσια νομικά που θα είναι ε, δεσμευτικά. Δεν θα μπορούμε δηλαδή διαρκώς να αναθέτουμε τις ελπίδες μας σε ιδανικές καταστάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η φωνή μας θα γίνει ακουστή και στην εξωτερική δράση. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική, σημαντικός ο πολιτικός διάλογος με τις χώρες που είναι υπό ανάπτυξη. Θα πρέπει να έχουμε διάλογο διαρκή με τις, ε, ε, την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει αυτά να συμπεριληφθούν κατά τη γνώμη μου στη γνωμοδότηση που ήδη είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Chair, and thank you to the... Uh, Κύριο Στία, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω και τον εισηγητή για την γνωμοδότηση που έχει προετοιμάσει. Είναι πολύ καλή βάση για συζήτηση. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι ξεκινά από την Ατζέντα 2030 που μόλις ε, υιοθετήθηκε καθώς επίσης και τους στόχους ε, ε, για την ανάπτυξη. Το κεφάλαιο που αναφέρεται στην καλή κυβέρνηση βεβαίως έχει ακολουθήσει και τις προηγούμενες μας ε, θέσεις ως Επιτροπή, το ίδιο και στον τομέα της σημασία που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για στην και συνεργασία. Θα ήθελα κάποιε διαφορές, ε, διαφορετήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, έναν οργανισμό που προωθεί ή υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, Promote or Defend. Σε αφορά τον τομέα της μετανάστευσης, χαίρομαι που γίνεται αναφορά σε αυτό το θέμα στην ονομαδότηση. Και σωστά λέει ο εισηγητής ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια απλοϊκή σκέψη ότι αν αυξήσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια θα μειωθούν οι μετανάστες που θέλουν να καταλήψουν τη χώρα τους. Στον τομέα της σχέσης των κόσμων των επιχειρήσεων με τα ανθρώπινα δικαιώματα πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το πρέπει να δείξουμε. Όπως είπε και η Μπεατρής φαντάζομαι αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της ε, συνάντησης των σκιωδών. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε εκεί. για θέματα τέτοιου τύπου είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές τους και όλους τους φορείς που τα επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω. Μέσω της διαδικασίας των τροπολογιών θα βελτιώσουμε, την, θα βελτιώσουμε ελπίζω τις ε, διατυπώσεις για παράδειγμα στη δεύτερη παράγραφο μια διορθώση που αφορά στην ε, ατζέντα την αναπτυξιακή στην οποία αναφερόμαστε. αυτέ είναι μικρέ διορθώσει που σίγουρα θα γίνουν. Κλείνω ευχαριστώντα τον εισηγητή για το εξαιρετικό κείμενο που έχει προετοιμάσει. Ωραία, ευχαριστούμε. Κύριο ε, όχι, λάθο, πριν σα δώσω το λόγο στην εισηγητή. Υπάρχει εκπρόσωπο του, όχι, δεν υπάρχει. Κύριο Φρούντζουλίτσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Και τον κύριο Πρέντα, αλλά και όλους τους άλλους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Πράγματι, πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τη σχέση που έχει η αναπτυξιακή συνεργασία και ο σεβασμός των ανθρωπινών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Επίσης, μάλλον θα έπρεπε να τονίσουμε περισσότερο τα θέματα της καλή διακυβέρνηση και τη καταπολέμησης της διαφθοράς. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί βελτιώνουν την ποιότητα της δημοκρατίας σε μια χώρα και να βελτιώσουν τον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί της. Πρέπει επίση να τονίσουμε το ρόλο που παίζουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και η κοινωνία των πολιτών, ο οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σε ορισμένε χώρε, όπου η διαφθορά είναι αυξημένη, τα προγράμματα της αναπτυξιακής συνεργασίας θα πρέπει να εφαρμόζονται, να υλοποιούνται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες αποδεδειγμένα να μπορούν να εξασφαλίσουν την διαφανή και ορθή χρήση των πόρων που θα τους στέλνουμε. Και πάλι ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ευχαριστώ να συζητήσουμε τις τροπολογίες που θα καταθέσετε. Ωραία, σας ευχαριστούμε να Σα ενημερώσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 19 Οκτωβρίου ε, τέλος της ημέρας και 10 Νοεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Έτσι ώστε μετά να, μετα... να το αποστείλουμε στην ΑΦΕΤ για την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο ε, θέμα της τη διάταξη. σημείο 13, προετοιμασία τη πρώτης παγκόσμια ανθρωπιστικής διασκέψη Κορυφή στην ε, Κωνσταντινούπολη. Είχαμε πρώτη Α, μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή που μας είπε πως εκείνη το προετοιμάζουν. Ο κύριος Σαλόμ, Σαλόμ, θα μας παρουσιάσει την ε, έκθεση του ως εισηγητής. Είναι η πρώτη τέτοια παγκόσμια διάσκεψη και πράγματι είναι ίσως και η πιο σημαντική στιγμή τώρα που ε, διοργανώνεται όταν έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ανθρωπιστική βοήθεια. Ενρίκε. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που σας ε, παρουσιάζω αυτή την έκθεση μετά από πολλές ώρες ε, επικοδομητικής εργασίας της Επιτροπής. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα ε, υπάρχει αυτή η, ένα τέταρτο του αιώνα υπάρχει αυτή η αναψηφιακή βοήθεια αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ο αριθμός των φυσικών καταστροφών έχει αυξηθεί με αναμφίβολα την επίπτωση των κλιματικών αλλαγών που είναι μια από τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Επίσης ε, οι ένοπλες σειράξεις έχουν ε, αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω του ότι υπάρχει ε, μεγαλύτερη ανασφάλεια ε, και οι φορείς που παρεμβαίνουν ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια έχουν επίσης αυξηθεί πολύ Υπάρχουν ε, πολλές ε, ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις για το περιβάλλον. Έχουν αλλάξει τα σενάρια όσον αφορά τους φορείς της ανθρωπιστικής βοήθειας επίσης, αλλά και υπάρχει και περιορισμός τελευταία των πόρων για την αντιμετώπιση των φυσικών ε, και ανθρωπιστικών καταστροφών, ιδιαίτερα μετά από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, η οποία μας ταλανίζει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ο ΙΕΣ, αυτό το πλαίσιο σε αυτό το σύνολο αλλαγών συγκαλεί την πρώτη ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφής ώστε να ε, ξανασκεφτούμε τη δομή του πλαισίου της ανθρωπιστικής δράσης και για να προσπαθήσει να συντονίσει αλλά και να καταφέρει να επιτύχει μεγαλύτερη συνοχή, αποτελεσματικότητα, συνεργασία στην απάντηση που θα δίνει στις ανάγκες των ανθρώπων, πράγμα που είναι ο απότερος στόχος και το ε, επίκεντρο της ανθρωπιστικής δράσης. Τη διάρκεια των τελευταίων μηνών και των τελευταίων ετών έχει, γίνει, έχει, έχει υπάρξει μια συμμετοχική διαδικασία μέσω της οποίας σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ανταλλάξει απόψεις, θέσεις για το πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το στόχο της επόμενης ανθρωπιστικής, της επερχόμενης μάλλον ανθρωπιστικής διάσκεψης κορυφής. Υπάρχουν όμως στοιχεία τα οποία δεν λειτουργούν όπως ήθιστε και μπορεί να περιορίσουν τον αντίκτυπο αυτής της διάσκεψης. Το βασικό είναι ότι δεν πρόκειται για μια διακυβερνητική διάσκεψη. Ε, αυτό σημαίνει ότι πολλές χώρες, ορισμένες εκ των οποίων παγκόσμιοι φορείς, δεν ε, δήλωσαν άμεσα συμμετοχή και δεν μάλλον συμμετείχαν άμεσα στην προετοιμασία αυτή τη διάσκεψης κορυφή. Ακριβώς επειδή δεν είναι διακυβερνητική διάσκεψη, η προπαρασκευή των εγγράφων, η δημιουργία αναζήτηση συμμαχιών και η, και η διαμόρφωση συνενέσεων είναι πιο περίπλοκη από ό,τι και από την ανθρωπιστική άποψη. επίση, μέχρι στιγμή δεν έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στις κρίσεις σε μακρά διαρκείες που είναι αυτές που αυτή τη στιγμή ε, απασχολούν τον περισσότερο κόσμο στην ε, στην Ιφίλιο και άρα απαιτούν ε, πιο δυναμική και έντονη ανθρωπιστική ε, βοήθεια. Πρόκειται λοιπόν για την ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφής που θα γίνει τον Μάιο τον επόμενο χρόνο στην Κωνσταντινούπολη και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιο σημαντική και βελτίωση. Καταρχήν ξεκινά μια διεθνής διαβούλευση ε, που ξεκινά στην Γενέβη την επόμενη εβδομάδα και έχουμε καλέσει την Ευρωπαϊκή Κομισιόν ώστε σε αυτή την παγκόσμια διαβούλευση να κρατήσει την πρωτοπορία, να κρατήσει ηγετική θέση, να προσπαθήσει να συνάψει ε, συμμαχίες και να εξέβρει συνενέσεις ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το νέο πλαίσιο Επίση, έχουμε προτάσεις που υπέβαλε η Προεδρία του Λουξεμβούργου, θα, θα υποβάλει συγγνώμη, στο τέλη του χρόνου ώστε το Συμβούλιο να υιοθετήσει ε, κάποιες θέσεις και να προωθήσει και τις θέσεις του προς τα κατημέλη και τέλος έχουμε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που προβλέπεται να είναι έτοιμη στις αρχές του επόμενου έτους και όπου ελπίζουμε πως θα έχουμε μια σαφή ε, πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτού του χρηματοδοτικού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν έχει ήδη ε, παρουσιάσει την ανακοίνωσή της που είναι πολύ θετική και την οποία εγώ ως συντάκτης αυτής της έκθεσης συμμερίζομαι πλήρως και που ε, όντως βρίσκει νέους τρόπους λειτουργίας ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή, η συνεργασία, να ε, εγγυηθεί την προβλεψιμότητα οικονομικής βοήθειας και ούτω καθεξής. Στην ανάπτυξη αυτής της θέσης λοιπόν που εκφράζει η Κομισιόν, η δική μου έκθεση ακολουθεί τρεις άξονες ε, ε, παγκόσμια κοινή δράση που προτείνω. Το πρώτο είναι το να προωθήσουμε δράσεις με γενική έννοια ανθρωπιστικής δράσης, στην οποία θα πρέπει να εξυπηρετεί και η Ευρωπαϊκή Συνένεση. Δηλαδή, το είπα ηθελημένο ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Συνένεση θα πρέπει να, να, αποτελέσει τη βάση γιατί δεν είναι εύκολο να προσπαθήσουμε να ε, ε, επιβάλλουμε τη δική μας δομή σε άλλους ε, διεθνείς φορείς αλλά μπορούμε να χρησιμεύσουμε ως παράδειγμα με τις καλές μας πρακτικές που μπορούμε να προσφέρουμε στους υπολείπους ώστε να μπορέσουμε από κοινού να προχωρήσουμε σε αυτή την παγκόσμια έννοια συνένεσης και ανθρωπιστικής δράσης σε πενταετή βάση ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε και να ανταποκριθούμε. Δεύτερος άξονας ο κώδικας διοντολογίας που θα βασίζεται στον σεβασμό των αρχών της ανθρωπιστικής δράσης και που θα επιτρέπει μεγαλύτερη συνοχή και συντονισμό. Σήμερα το πρωί, όπως έλεγε και η Λίντα ε, και ο Λεφλε ω εκπρόσωπο τη Υπηρεσία Εξωτερική δράση τόνιζαν διαρκώ πόσο πολύ ο συντονισμό του συντονισμού ω συντονισμέ είναι βασική, ε, ε, το βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να διέπει κάθε ανθρωπιστική δράση. Ε, έτσι ώστε να σεβόμαστε αυτές τις κοινωνίες τις οποίες θέλουμε να βοηθήσουμε τους ε, απολύτες τους που βρίσκονται σε κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης. Ανθρωπιστική δράση λοιπόν, εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν επιθυμώ, ούτε πιστεύω πως ε, θέλουμε εμεί ως Επιτροπή ή ως Κοινοβούλιο ε, να ζητήσω κάποιο ακόμα χρηματοδοτικό μέσο, γιατί όταν μιλώ για παγκόσμιο ταμείο, εγώ είμαι έτοιμος να δεχτώ να συγχωνευτούν τα κονδύλια που ήδη υπάρχουν ώστε να λειτουργήσουν ίσως καλύτερα. Να... Και ε, η Λίντα το είπε ότι ήδη πολύ συχνά μπερδευόμαστε να παρακολουθήσουμε πόσα ταμεία, πόσες ε, ε, ΜΚΟ, πόσοι συγκεκριμένοι φορείς λειτουργούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης, προβλεψιμότητα δηλαδή της χρηματοδότησης, να γίνεται όσο δίνεται ε, καλύτερη χρήση των όσων έχουμε στη διάθεσή μας και άρα αν τελικά, ναι, πούμε ότι ναι, φτιάχνουμε ένα παγκόσμιο ταμείο ε, στην Ισταμπούλ, στην Κωνσταντινούπολη, να αποτελέσουν όλα αυτά μέσω, το ίδιο μέσο, την ίδια ροή τη χρηματοδοτική για την αντιμετώπιση των αναγκών. Στην έκθεσή μου θα βρείτε την επιβεβαίωση των αρχών της ανθρωπιστικής δράσης. Αυτό είναι ένα στοιχείο που είναι κάτι που ζητούν όλοι οι ανθρωπιστικοί φορείς, θα δείτε και το επίκεντρο, το επίκεντρο προς τους ανθρώπους που, απε... που, που, χρήζουν βοήθειας, όλα τα υπόλοιπα είναι... Ε, τα, ε, παρα, οι παράπλευρες ε, προσπάθειες ώστε όντως να βοηθήσουμε όλους αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Μιλάμε για την ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά θα δείτε πως υπάρχει και μία πτυχή ενίσχυση των τοπικών φορέων, μία πτυχή που ακολουθεί πως το γεγονό ότι συχνά επιτόπου οι τοπικοί φορείς που δρούν εκεί δηλαδή τόσο της κοινωνίας εκεί όπου δηλαδή βοηθάμε, όπως ας πούμε και οι φορείς που είναι οι μη κυβερνητικοί, οι διεθνείς φορείς, είναι αυτοί επιτόπου οι άνθρωποι που πρέπει και οφείλουν να βοηθήσουν και να ε, αναπτύξουν και να, μάλλον, να συμπεριφερθούν με βάση με αυτές τις αξίες. συνεργασία είχα με την ΕΚΟ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Αντιπρόεδρο Γεωργέβα, που προετοιμάζει την ευρωπαϊκή θέση σε σχέση με το πάνελ υψηλού επίπεδου για την χρηματοδότηση Προετοιμάσαμε και μια σειρά τροπολογιών, περισσότερες από αυτές τονίζουν μια κλειδιά όπως η προστασία των ε, ομάδων ε, κινδύνου, την προστασία των, ε, εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια που όλο ένα και περισσότερο ρισκάρουν τη ζωή τους και πολλές φορές την χάνουν σε πολύ μεγάλα νούμερα ενώ προσπαθούν να βοηθήσουν σε ανθρωπιστικές κρίσεις, ε, επίση προτάσεις ε, χρηματοδότησης που κατευθύνονται προς τους τοπικούς φορείς, καθώς και ένα πολιτικό πλαίσιο δράσης, ε, μάλλον ένα πλαίσιο πολιτικής δράσης για τα κράτη τα οποία έχουν καταρρεύσει, μια αναπέτηση προς τους δωρητές για μεγαλύτερη ευελιξία, επαγγελματισμό και διαφάνεια, καθώς και μια αποδοχή για την ιδιωτική συμμετοχή από τη στιγμή που αυτή βασίζεται στο σεβασμό και στην εφαρμογή των ανθρωπιστικών αρχών. Γίνεται επίση μια αμνία στη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας κάτι ακόμα που, ήδη που ανέφερα ήδη. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Συνένεση θα πρέπει να ενισχύσει τη θέση μας, χωρίς να προσπαθήσει όμως να την επιβάλλει σε οποιονδήποτε, ούτε καν να προσπαθήσουμε να την παρουσιάσουμε στην καλύτερη δυνατή λύση, αλλά να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι στο δικό μας πλαίσιο το η ευρωπαϊκή προσπάθεια δίνει καλά αποτελέσματα και άρα αν έχουμε μια παγκόσμια συνένεση με κοινέ αρχές θα μπορούσε να βοηθήσει στο να λειτουργήσουν τα πράγματα ακόμη καλύτερα στο μέλλον. Και θα κλείσω ευχαριστώντας ε, κυρίως την Ενρίκα που συνέβαλε στην εργασία διαδικασία που η έκθεσή μου χωρίς τη βοήθεια αυτή δεν θα ήταν τόσο καλή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Ρίκια. Ο κύριος Γκέρεντς. Α, συγγνώμη. Σαν και μετά θα ακούσουμε τον άλλο. Και εγώ θέλω να μιλήσω. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο του φίλου μου του Σαλομγερέρο. Είναι πολύ πλήρης η έκθεσή του. Και είναι πολύ σημαντικά τα θέματα που αναδεικνύει. Και εντυπωσιακή έκταση επίσης η έκθεση. τελικά η αιτιολογική ήταν μικρότερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει καταλήγει να αναδεικνύει τα σημαντικότερα θέματα αυτά που θα έπρεπε να αναδείξει η Επιτροπή μας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε γιατί καταλήγουμε σε αυτή την διάσκεψη η οποία είναι μια συμβουλευτική διαδικασία. Δεν είναι διακυβερνητική διάσκεψη το οποίο είναι θετικό, γιατί σημαίνει ότι αυτή η συμμετοχή ε, έχουμε δει ότι η συμμετοχή ε, άλλων φορέων εκτός των κυβερνήσεων, αυτή η πολυμερής προσέγγιση λειτουργεί. Το είδαμε και στην Αντισάμπαμπα. Είναι ευχάριστο λοιπόν το γεγονό ότι αυτή η πολυμερή προσέγγιση δεν κινδυνεύει τόσο πολύ πια. Αναφέρεται η σημασία του επαγγελματισμού που πρέπει να ε, έχουν οι εκείνοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα τη ανθρωπιστική βοήθεια και επειδή ακριβώ έχουν την ιδιαίτερη γνώση του τι συμβαίνει επί τόπου, επειδή βρίσκονται επί τόπου, μπορεί να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια. Το είδαμε για παράδειγμα στην κρίση του ιού του έμπολα, ε, στη συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό ή με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, είδαμε πόσο μεγάλη σημασία είχε το γεγονό ότι μπορούσαν να ενημερώσουν και τον τοπικό πληθυσμό. Βρίσκονταν έτη φωτός ε, πιο μπροστά από, για παράδειγμα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. η ανθρωπιστική βοήθεια έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι εντυπωσιακή τις πρώτες τρεις ημέρες όταν ξεσπάει η κρίση που έχει τεράστια δημοσιότητα και το διαπιστώνουμε επίσης αυτό και στη χρηματοδότηση. Οι δωρεές αυξάνονται με τεράστιους ρυθμούς τις πρώτες μέρες και μετά πέφτουν. Και καταλήγουμε με πολλές ξεχασμένες κρίσεις. λοιπόν η αποκέντρωση και η απόδοση ευθυνών περισσότερων στους τοπικούς φορείς λειτουργεί σωστά. Στο Τσάντ, έχω ένα άλλο παράδειγμα, η υπηρεσία του ΟΗΕ που βρίσκεται εκεί, α, μάλλον η, η, ε, το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα αυτών. Στην Κουντούζ, οι γιατροί των γιατρών χωρίς σύνορα και οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο εκεί δολοφονήθηκαν. Δεν μπορεί κατά κανέναν τρόπο να δικαιολογηθεί αυτή η επίθεση. γεγονό ότι το νοσοκομείο βρισκόταν εκεί ήταν απολύτω γνωστό σε όλε τι δυνάμει που ήταν παρούσε στο Αφγανιστάν, επομένω είναι απολύτω απαράδεκτο αυτό που έγινε. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε ω κοινοβούλιο αυτό που συνέβη στην Κουντούζ. Θα πρέπει να απαιτήσουμε λογοδοσία, θα πρέπει να απαιτήσουμε επίση αποζημίωση των θυμάτων, αλλά και λογοδοσία προ τη διεθνή κοινότητα και προ την κοινότητα εκείνων των ανθρώπων που συνεισφέρουν στι ανθρωπιστικέ ε, επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα τους γιατρούς χωρίς σύνορα, που ξέρουμε τι θυσιάζουν σε αυτές τις αποστολές. Οφείλει κατά την άποψή μου λοιπόν, να, να λάβει ε, θέση και να πει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκάθαρα ότι ήταν απαράδεκτο αυτό που συνέβη στην Κοντούς. Πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να τεθεί στην επόμενη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως θέμα. αυτά από την πλευρά μου με όλες τα, τα συγχαρητήρια που αξίζει ο συνάδελφος Γεραίρο. Πιστεύω. Α, ξέχασα κάτι. Ένα τελευταίο σημείο. Το ζήτημα της χρηματοδότησης. Εδώ και πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμαρτύρεται για την έλλειψη πόρων. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωπή κονδύλια που κανονικά είχαν προγραμματιστεί για επόμενες χρονιές. Περιμένω μια χρηματοδότηση του ε, προγραμματίζουν μια χρηματοδότηση του ύψους των 4 δισεκατομμυρίων και φτάνουμε στο 1 Το οποίο σημαίνει ότι απλώς δίνουμε υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται στην πράξη. αυτή η συζήτηση για τη χρηματοδότηση μου θυμίζει τον έξοδο που κάποιος είχε, καλέσει, είχε προετοιμάσει φαγητό για πέντε άτομα, ήρθαν δέκα, αλλά στο τέλος πάλι, κάτι έμεινε, δεν το φάγαν όλα, γιατί όλοι ήθελαν να είναι ευγενικοί, επομένως πάντα βρίσκουμε δικαιολογίες. Αλλά για να είμαστε ειλικρινεί, δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι. Δεν έχουν προ... προπολογιστεί αρκετοί πόροι. το 0,7% του ΑΕΠ. Εάν είχε τηρήσει αυτήν την δέσμευση της Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων στην Αφρική. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και έχουμε τον κύριο Στήρ τώρα. Και θα τον κύριο Κουλογλού. Ο κύριος Στήρ πρώτος όμως. Ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σας Ρίκε για την εξαιρετική έκθεση, το σχέδιο έκθεσης που μας παρουσίασε. Τα διάβασα στα κροατικά, θα συνεχίσω λοιπόν στα κροατικά. Έχω την εντύπωση ότι το έγγραφο αυτό είναι πραγματικά εξαιρετική σημασία, δεδομένη και της πολιτικής ορμής που θα υπάρχει και που θα δοθεί και στην επόμενη ολομέλεια που θα συζητήσουμε το θέμα. Όσοι συμμετείχαμε στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Νέα Υόρκη, όπου τέθηκε το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάπτυξη, μπόρεσαν να δουν με, από πρώτο χέρι την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν ε, υπό επίθεση για την ανθρωπιστική κρίση, για την προσφυγικό. Νομίζω ότι η επικέντρωση λοιπόν του Ενρίκε στην μετάβαση από μία θέση άμυνας σε μία θέση ισχύως προκειμένου να επανατοποθετήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, ικανή και ηγετική στα ζητήματα αυτά αποτελεί τη σωστή προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πρέπει να αντιληφθούμε και την διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης που θα λάβει χώρα το επόμενο έτος του χρόνου. Αλλά αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι όντως μιλάμε για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημείο αυτό. Και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή με τον τρόπο που προβλήθηκε είναι πάρα πολύ επίκαιρη και πάρα πολύ εύστοχη. Έτσι θα πρέπει να δράσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό ορίζεται στην τρίτη παράγραφο. Όπου προτείνεται ένα πενταετές πρόγραμμα και ένα follow-up των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Αυτό δεν αποτελεί μια γενική, γενικευμένη θέση. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε προτάσει που περιλαμβάνονται το θέμα του συντονισμού. Προφανώ στο διεθνέ προσκήνιο, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη το μορφότυπο τη ε, διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και αυτό λοιπόν θα αποτελέσει άλλη μια πρόκληση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε άλλο ένα στοιχείο. Και το τονίζει μάλιστα η έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κυρέρο γιατί στην ενδέκατη η παράγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αύξηση ενδεχομένως του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις κρίσης από 2-4%. Το συζητήσαμε αυτό και χθε, αλλά το γεγονό ότι έχει μπει και στο σημερινό έγγραφο είναι σημαντικό και ήθελα να το υπογραμμίσω. Ευχαριστώ λοιπόν τον ε, Ενρίκε που τα συμπεριέλαβε όλα αυτά στην εκθέση του. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πρόεδρο. Η κυρία Μπεσέρα. Και συνάδελφοι, δεν έχουμε. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, ο κύριο Κούλογλου. Πολύ λυπάμαι. Εγώ έκανα λάθο. Έχουμε. Έχουμε και την ερώτησή σου προ την Επιτροπή, Ενρίκε. Έχετε το λόγο. Δηλαδή, no, you first. No, no, no, no. Αν είναι η γυναίκα... Όχι, όχι, εσείς πρώτος. Women ε, first, if you like. No, no, it's fine. You, you go ahead because be waiting. Όχι, όχι, εσείς, εσείς γιατί περιμένετε ώρα. Και μετά η Μπέτρης. Ωραία. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό και εύστοχο σχέδιο από τον συνάδελφο Ερίκε Γκερέρο. Δεν θέλω να επαναλάβω πολλά πράγματα υπάρχει μια εκτόπιση πληθυσμών σήμερα, μετακίνηση πληθυσμών προσφύγων που είναι μεγαλύτερη από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ειδικότερα στην ε, περιοχή όπου, από όπου προέρχομαι εγώ και στη χώρα, στην Ελλάδα, το βλέπουμε καθημερινά. Και σε μεγάλη έκταση, σε δραματική μορφή. Και φοβάμαι ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία ε, με την ε, με τις πολύ δολοφονικές ε, βοβιστικές επιθέσεις θα προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση και στην Τουρκία και σε όλη την περιοχή και στην ε, Συρία. Η Τουρκία ενδεχομένως να μην μπορέσει να λειτουργήσει σαν ο τόπος παραμονής των προσφύγων όπως ε, σχεδίαζαν και το είδαμε με τις ομιλίες του της προηγούμενης εβδομάδας και ο κύριος Ολάντ και η κυρία Μέρκελ. Αυτό ίσως δεν θα μπορέσει να γίνει και πρέπει ίσως συνάδελφοι να προετοιμαζόμαστε για μεγαλύτερα κύματα προσφύγων και από αυτά που έχουμε ήδη δει αυτόν τον καιρό. Για πολλές χώρες, όπως και για τη δική μου, η κατάσταση είναι πλέον πέρα από τις δυνάμεις μας και πρέπει κάποια στιγμή πιστεύουμε να αρχίσουμε να μιλάμε και για τα αίτια που γέννησαν όλες αυτές τις καταστροφές. Και γι' αυτό σκοπεύω να καταθέσω σχετική τροπολογία. Ένα άλλο σημείο ε, είναι το μιλώντας για τα αίτια και μιλώντας για τις δυνάμεις εκείνες που δημιούργησαν με τη δράση τους τα, ε, αυτά τα μεγάλα κύματα προσφύγων από το Ιράκ, ε, από τη Συρία, από το Αφγανιστάν είναι το περιστατικό που έγινε στην Κουντούς με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου των γιατρών χωρίς σύνορα. Υποστηρίζω έθερμα την ε, πρόταση του συναδέλφου Γκέρενς που μόλις έκανε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε συζητήσει και μία έρευνα για το, τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτό το έγκλημα, ενώ αυτοί οι οποίοι βομβάρδιζαν γνώριζαν πολύ καλά ότι επρόκειτο για νοσοκομείο, το οποίο μάλιστα σε διάστημα μίας ώρας δέχτηκε επανειλημμένες βομβιστικές επιθέσεις. Ένα ακόμα σημείο είναι φυσικά η επιπτώση της κλιματικής αλλαγής, και οι κλιματικοί πρόσφυγες, οι πρόσφυγες από την αλλαγή του κλίματος που περιμένουμε. Και εδώ θα ήθελα να καταθέσω, επιφυλάσσουμε να καταθέσω μια τροπολογία για αυτό το θέμα. Ένα τελευταίο σημείο είναι για την προστασία των προσφύγων και αυτών που έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς που πρέπει και αυτοί να, έχουν, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτισμικές, και θρησκευτικέ επιλογές που έχουν. Παραδείγματο χάρη το δικαίωμα στην έκτρωση που απαγορεύεται ρητά από ορισμένε θρησκείε πρέπει στους χώρους υποδοχής των προσφύγων να, ε, να γίνει απόλυτα σεβαστό σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά τον συνάδελφο για την ε, εξαιρετική δουλειά και εσάς που με ακούσατε. Um, thank, thank you very much. Now, so now it's Beatrice Becerra and then Heidi Hautila. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, συνάδελφοι, μέχρι τις 5.30 γιατί μετά έχουμε την κοινή ε, συνεδρίαση με ε, την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Γεωργίας. Πεατρίς, όσο πιο γρήγορα απολύτω. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω μόνο να κάνω μια αναφορά στον κύριο ε, Γερέρο, εκτό από το να τον ευχαριστήσω για το ε, τεράστιο έργο του. Ε, θα λαβεί υπόψη και η νομοδότηση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είναι πολύ καλό που η Λένα Βαλεντιάνο θα είναι εισηγήτρια στην Επιτροπή της ΑΦΕΤ ε, και πιστεύουμε ότι αυτή η δέσμευση ε, σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σημαντική για τον στόχο τον οποίο ε, θέλουμε να επιτύχουμε, δηλαδή να βελτιωθεί η χορήγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα ήθελα μόνο να τονίσω τα όσα θα Ελπίζω να ληφθούν υπόψη κάποιες στοιχές όπως ας πούμε το δικαίωμα της ε, πρόσβασης στο νερό αλλά και ένα ανθρώπινο δικαίωμα που είναι θεμελιώδες και που συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα στη ζωή και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης, η διεθνής ε, ανθρωπιστική νομοθεσία καθιστά το δικαίωμα στην πρόσβαση ενός μεγάλου στην πρόσβαση σε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών ε, ε, αναπαραγωγικής υγείας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται μέσα στην ανθρωπιστική ε, βοήθεια. Θα πρέπει να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί αυτή η σχέση, η η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στη δημοκρατία και την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πυροπαρασκευή αυτή τη διάσκεψη κορυφή. Ευχαριστώ, Χαϊδη. Να προσθέσω και εγώ μερικέ παρατηρήσει από πλευρά τη ομάδα μου. Καταρχά, καλωσορίζουμε τέρο του σχέδιου έκθεση του συναδέλφου Γκερέρο Σαλόμ και τι τροπολογίε που υπέβαλε. Θεωρούμε ότι μπορούμε να τι υποστηρίξουμε. Να αναφέρω εν συντομία τα θέματα τα οποία θεωρούμε την εξαιρετικά στο σχέδιο έκθεση. Καταρχά, η επικέντρωση στι ευαίσθητε ομάδε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, γιατί πολύ συχνά οι ανάπηροι, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκε βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στι ανάγκε του. Επίση, κατά δεύτερον, η προσέγγιση βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία αυτών. Κατά τρίτον, η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή υποστήριξης στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη. Συμφωνούμε για όσα αναφέρονται για τη διαφάνεια, την πρόσβαση και σε πολλές περιπτώσεις, όπως ξέρετε, υπάρχουν ε, εντόνωτα προβλήματα από την Ουκρανία και στο κενό στη χρηματοδότηση, το οποίο το συζητήσαμε και χθες Επίσης, να επενθυμίσουμε και την ανάγκη αντιμετώπισης των βασικών αιτιών των κρίσεων. Τι θα θέλαμε να προσθέσουμε τώρα. Να τονίσουμε μία προσέγγιση βάσει του φίλου πιο πολύ. Να αναφερθούμε πιο έντονα στην κλιματική αλλαγή και στις ξεχασμένες κρίσεις που δεν ε, συγκεντρώνουν την προσοχή του κοινού απαραίτητο. Να πούμε δύο λόγια παραπάνω και στις εκτοπισμένα άτομα στις χώρες υποδοχή. Ο ρόλο των ΜΚΟ στην ε, παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη επίση μα απασχολεί. Δεν θα ακρηγορήσω. Ευχαριστώ τον εισηγητή και προσβλέπω στην ε, καλή συνεργασία για την επιτεύξη ενό υψηλού επίπεδου συμβιβασμού. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Δύο σημεία από πλευρά μου εδώ και θα ήθελα να αναφέρω. Χθε, όταν συζητήσαμε το θέμα τη εκπαίδευση για τα παιδιά σε καταστάσει εκτάκτου ανάγκη και σε παρακαταμένε καταστάσει, το 4% αναρωτιέμαι είναι αρκετό. Από την Επιτροπή κάποιοι μας είπαν ότι μπορεί και να μην αρκεί. Μήπως θα πρέπει να βγούμε τουλάχιστον 4% γιατί όσο πιο πολλές οι κρίσεις, τόσο και πιο, πολύ, πιο πολλές, πολλές οι ανάγκες. Εξαρτάται από τον προπολογισμό φυσικά. Ύστερα. Και πολλοί συνάδελφοι το ανέφεραν αυτό με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, την επίθεση στα νοσοκομεία. Μήπως θα μπορούσαμε να θέσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια των ε, καταστάσεων αυτών, γιατί ακούσαμε χθε ότι είναι όλο και πιο δύσκολο για τα άτομα αυτά να πάνε στη δουλειά του. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε και να τηλεφκάνουμε τι έγινε ακριβώ. Και είχαμε και ανάλογε περιστάσει, περιπτώσει στη Γάζα με βομβαρδισμό νοσοκομείων για την προστασία του εργατικού δυναμικού δηλαδή. Γιατί άλλο δεν θα μείνει κανένα. Για να βοηθάει στι δύσκολε καταστάσει η κυρία Λενιονέτο, διευθύντρια από την ΕΚΟ. Αν θέλετε να κάνετε δύο σχόλια. δεν έχουμε πολύ χρόνο, πολύ λυπάμαι που σας πιέζω, αλλά αν θέλετε να είστε σύντομοι. Thank you, Chair. Just very briefly, the Commission... Σας ευχαριστώ. Από την πλευρά της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννα Ροσαλόμ. Είναι πολύ χρήσιμη η έκθεση που έχει προετοιμάσει και ταιριάζει και με την ανακοίνωση που έχει προετοιμάσει η Επιτροπή προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αναφέρει ο κ. Χερέρο στην εισαγωγή της εκθεσής του, ε, αναφερόμενοι στις αρχές που θα πρέπει να γίνονται ε, να σεβαστές κατά τη διάρκεια της παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα ήθελα επίσης να σας βεβαιώσω ότι και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να εργάζονται στον τομέα αυτό για την προετοιμασία δηλαδή της πρώτης παγκόσμιας ανθρωπιστικής διάσκεψης. Ε, έχει προετοιμαστεί ότι ε, έχει υπάρξει μια συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα δημοσιοποίησε τη θέση, την κοινή των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπέρους δηλαδή της Ένωσης. Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει τις θέσεις που καταγράφονται στην έκθεση του κ. Σαλόμ. Και στην ανακοίνωσή μας αναφέραμε ότι αυτή η διάσκεψη είναι μια ευκαιρία για να επαναβεβαιωθούν οι βασικές αρχές την παροχή της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Και όπως είπε και ο κύριος Γεράρος Σαλόμ, πράγματι αυξάνονται οι ανάγκες και δεν αυξάνεται με αντίστοιχους ρυθμούς δεν αυξάνονται με διαθέσιμους ρυθμούς ε, διαθέσιμοι πόροι, οι προπολογισμοί. Ίσως ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι ένα παγκόσμιο ταμείο. Όπως είπε και ο κύριος ε, Σαλόμ, η Επίτροπος Γεωργίευα θα προεδρεύσει του πάνελ υψηλού επίπεδου για τη χρηματοδότηση. Θα αναμείνουμε τα αποτελέσματα αυτού του πάνελ. Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει παράλληλα να εργαστούμε και στο ζήτημα της αποτελεσματικότητας και της χρηματοδότησης, της εξέβρισης των πόρων. Έχουμε και εμεί την ε, ανακοίνωσή να αναφερθεί στη σημασία της αποτελεσματικότητα τη χρήση αυτών των πόρων. Αυτά από την πλευρά μου. ευχαριστώ. Εμεί σα ευχαριστούμε. Ενρίκε. Μάλιστα, θα είμαστε γίνεται πιο σύντομο. Έχω σημειώσει και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφου για τι ε, συμβολές τους. Πιστεύω πως υπάρχει μεγάλος βαθμός συνένεσης ε, στο ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο την προστασία των ε, ανθρωπιστικών φορέων ε, και στον συντονισμό τους καθώς πρόκειται για διάσκεψη κορυφής που δεν είναι διακυβερνητική όπως και για τις κλιματικές αλλαγές, να τονίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προπτική του φύλου, την αντιμετώπιση των ξεχασμένων κρίσεων, την ασφάλεια και την προστασία των ανθρωπιστικών φορέων. Ένα-δυο σχόλια έχω να κάνω μόνο που πιστεύω πως είναι σημαντικό από την αρχή να ε, είναι ξεκάθαρο. Ε, Καταρχήν πρόκειται για διάσκεψη κορυφής που θα γίνει στην ε, Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτό θα πρέπει να συγχαίρεται με την κατάσταση ε, στην Τουρκία. Αυτή είναι μια διάσκεψη κορυφής στο ΙΕ που συγκαλείται στην ε, Κωνσταντινούπολη που θα μπορούσε να συγκληθεί και στην Μαδρίτη. Οπότε τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία, την κατάσταση στην Τουρκία κτλ. κτλ θα πρέπει να ε, μην έχουν, μάλλον δεν έχουν χώρο σε αυτήν εδώ την έκθεση. Έπειτα η ευρωπαϊκή κρίση που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη δική μας θέση σε αυτήν την ε, διάσκεψη κορυφής. Γιατί Όσο καλύτερα ανταποκρινόμαστε, θα έχουμε και μεγαλύτερη ηθική δύναμη. Ε, και το αντίστροφο ισχύει όμως. Δεν θα αποτελέσουμε παράδειγμα για κανέναν, εάν δεν ε, να αντιμετωπίσουμε σωστά. Πάντως, δεν μπορούμε να πάμε στην Κωνσταντινούπολη για να τονίσουμε ε, τη δική μας ανθρωπιστική κρίση, γιατί για ολόκληρο τον κόσμο αυτή η κρίση που εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει σε ένα σωρό μέρη. Στην από Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, εκτοπισμοί πληθυσμών, μετακινήσεις πληθυσμών, δηλαδή να μην στρέψουμε την προσοχή σε εμά, να μην χαρακτηριστούμε ως εγωκεντρικοί, ε, δηλαδή λες και το δικό μας πρόβλημα είναι το σημαντικότερο, ενώ πολλές φορές τα προβλήματα των υπολείπων είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που έχουμε εμείς. Νομίζω λοιπόν πως ε, είναι, ε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να αναφερθούν, αλλά να ξεφύγουμε από την ε, εγωκεντρική ευρωπαϊκή θέση, ενώ συμμετέχουμε σε μια διεθνή διάσκεψη κορυφής, την οποία έχουν συγκαλέσει τα ενωμένα Έθνη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το κουντούς η κουντούς Συζητήθηκε, ήμουν στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Συζητήθηκε και θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και αυτή η υπόθεση και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να ε, υπάρχει μια εξήγηση για το τι συνέβη στην Κουντούς γιατί δυστυχώς θα γίνει ξανά στο μέλλον. Αλλά στο βαθμό που εμείς θα έχουμε υψώσει τη φωνή μας κατά τέτοιων γεγονότων και ε, θα είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που υπάρχουν ε, στοιχεία ε, γιατί ανθρωπιστικοί φορείς δεν θα πρέπει να αισθάνονται φρένο επειδή λειτουργούν σε πλαίσιο σύγκρουσης και πόλεμης σύραξης. Την Δευτέρα στις 5 θα μιλήσουμε ξανά για αυτήν την έκθεση. Παρακαλώ συζητήστε με τον Ερίκε αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο μας, ε, η ώρα των ε, ερωτήσεων θα αναβληθεί γιατί ήταν η ερώτηση του κ. Γκερέρο και συμφώνησε να αναβληθεί για την επόμενη μας συνεδρία. Σε αναβάλλεται το 15-16 στα διάφορα. Έχει κανείς κάτι να συζητήσουμε στα διάφορα? Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημείο 17. Επόμενη συνεδρίαση. προγραμματισμένη συνεδρίαση επόμενη είναι στις 9 ε, Νοεμβρίου το απόγευμα και την επόμενη μέρα, ε, όλη την ημέρα. Και έχουμε και δύο έκτακτες. Μία την 5η το πρωί στις 9 μαζί με την ΑΦΕΤ. Φαντάζομαι ότι είναι για την Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για τη ψηφοφορία για το βραβείο Ζαχάροφ του 2015 και έπειτα στις 9 Οκτωβρίου, δηλαδή μια 19, σε μια εβδομάδα δηλαδή, ειδική έκτακτη συνεδρίαση με τον Επίτροπο Μίμητσα. Δύο έκτακτες λοιπόν συνεδριάσεις. Και τώρα συνάδελφοι, έχουμε αμέσως τώρα κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Γεωργίας για μια ώρα για να ε, μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα ε, διατροφής, τροφίμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα πάμε στην 3 σε 50 απέναντι την Ολομέλεια.